Uh, λοιπόν, έφτασε η ώρα να ξεκινήσουμε με τα θέματα που έχουν απομείνει στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο είναι το υπαριθμό 7. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού της Οικονομικής Πολιτικής. Η εισηγήτρια είναι η Περβάνς οπότε έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θελήσατε η Επιτροπή μας να συντάξει έκθεση πρωτοβουλία για το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ε, όχι μόνο για τη δική μας Επιτροπή, αλλά και για το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι σημαντική υπόθεση. Η προσέγγιση ε, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής η αφετηρία που επέλεξε για να αρχίσει τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση καταλήγει στις έξι εκθέσεις ε, που και η Επιτροπή μας ε, θα λάβει γνώση και θα αποφανθεί. Η παρούσα λοιπόν έκθεση πρωτοβουλίας στο παρόν στάδιο δεν έχει ως στόχο να είναι έκθεση επί της ουσίας ε, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αλλά ένα πλαίσιο αναφοράς και μόνο, βάσει του οποίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τα επόμενα χρόνια θα έχει ακριβώς ένα μπούσουλα για να ασχοληθεί με το περιεχόμενο και την ουσία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επίσης, σκοπός της έκθεσης αυτής δεν είναι να ε, επισέλθει σε θέματα των έξι εκθέσεων για την οικονομική διακυβέρνηση, των οποίων θα λάβετε γνώση. Αλλά όλες αυτές φυσικά οι εκθέσεις θα ενταχθούν ε, στο αρχιτεκτόνημα αυτό που αυτή τη στιγμή οικοδομούμε. Πέρα λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σκοπό και στόχο να καθορίσει τις προϋποθέσεις και τους όρους εκείνους βάσει των οποίων μπορεί να οργανωθεί η πολιτική συζήτηση. Γιατί όταν μιλούμε για οικονομική διακυβέρνηση δεν ε, εννοούμε φυσικά μόνο τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε. Γίνονται επιλογές για τις οικονομικές πολιτικές που θα ακολουθηθούν. Και το θέμα της οικονομικής λειτουργίας τίθεται με τρόπο πάρα πολύ κομβικό και κρίσιμο. Euh, η δημοκρατία θα πρέπει να έχει σημαντική ύπαρξη σε αυτό το εξάμεινο και λόγο. Άρα ε, η διασύνδεση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εθνικών Κοινοβουλίων είναι σημαντικό στοιχείο. Αλλά και κάτι ακόμα, ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων. Γνωρίζουμε τώρα ότι οι κοινωνικοί εταίροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετέχουν σε μια άσκηση που ονομάζεται μακροοικονομικός διάλογος. Αλλά μέχρι σήμερα εμφανίζεται ως πάρα πολύ τυπικός διάλογος. Για το περιεχόμενο τώρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Κοιτάζοντας τις έξι εκθέσεις που συζητούμε σήμερα, μου έκανε εντύπωση και με ενσύχησε κάτι. Όλες αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε γύρω από την έννοια της οικονομικής διακυβέρνησης, οφείλουν την ύπαρξή τους ε, στην εξή κατάσταση. Έχουμε μια, οικονομική, μια νομισματική ένωση που από την αρχή λειτουργεί με τρόπο ομοσπονδιακό και μια οικονομική πολιτική που ασκείται από τα κράτη-μέλη και μια προσέγγιση γεννού ενδιαφέροντος βάσει το άρθρο 121 της συνθήκης. Αυτό που στην αρχή λοιπόν ήταν ε, ένα ζήτημα ε, συντονισμού αμυγός, σήμερα εμφανίζεται ως ένα ε, θέμα εποπτείας και κυρώσεων αποκλειστικά. Μα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει οικονομική πολιτική που να είναι μόνο εποπτεία. Το διακύβευμα εκεί και το ζητούμενο είναι πρώτα απ' όλα ο συντονισμός όχι ο συντονισμός της εποπτείας και των κυρώσεων, αλλά ο συντονισμός της εκτίμησης των καταστάσεων και ο συντονισμός του τι πρέπει να κάνουμε και καλώ τους εισηγητές του πακέτου της οικονομικής διακυβέρνησης να χτενίσουν τα κείμενα και να βάλουν και λίγο συντονισμό σε αυτά και να μην αναφέρεται μόνο η εποπτεία. Ξέρω εγώ βάλετε συντονισμό και εποπτεία, αλλά μην χαθεί τελείως ο συντονισμός, διότι διαφορετικά δεν κάνουμε τίποτα. Ωραία, εποπτεύουμε, επιτηρούμε και συνέχεια μαστιγώνουμε και πίπτει ράβδος. Και λοιπόν έτσι θα πετύχουμε την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Δεύτερη σημειολογική παρατήρηση. Τι ε, είναι αυτό το εγχείρημα που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Στη νομισματική πολιτική έχουμε δύο περιορισμούς. Πρώτον, είναι πάρα πολύ ε, ομοσπονδιακός ο χαρακτήρας της από τη μια και από την άλλη πρέπει πλήρως να ενταχθεί στο σεβασμό της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας. Ακριβώς επειδή είναι ανεξάρτητη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κανείς δεν επιθυμεί να αμφισβητήσει αυτό το καθεστώς της, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, θα θυμούνται μερικοί, ο κύριος Γκασία Μαργκάγιο, γιατί ήδη ήταν ε, μαζί μου μέλος, το είχαμε πει όταν εφήβραμε την έννοια του νομισματικού διαλόγου. Γιατί το κάναμε αυτό. Γιατί δεν μπορούσαμε να ελέγχουμε την Κεντρική Τράπεζα διότι είναι ανεξάρτητη. Δεν μπορούμε λοιπόν πλήρως να μεταφέρουμε ε, την έννοια του διαλόγου στο μακροοικονομικό πεδίο, διότι υπάρχουν οι μεγάλοι προσανατολισμοί οικονομικοί ε, και πολιτικοί και ε, προσανατολισμοί για την απασχόληση. Με όλα αυτά ασχολούμαστε, αλλά προς Θεού μην ενοχλήσουμε στην ανεξαρτησία της στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βέβαια, εγώ δεν είμαι συμφωνία απολύτως με αυτό το πνεύμα ε, και σας παρακαλώ ε, να το σκεφτούμε λίγο, να συνεργαστούμε, να brainstorming για να βρούμε τη σωστή προσέγγιση. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα, τα γνωρίζετε όλοι πολύ καλά. Αρχίζει ο κύκλος με την αρχική εξέταση της ανάπτυξης για τις οικονομίες με τα τρία παραδείγματα, στρατηγική 2020, μακροοικονομική πολιτική και έκθεση για την απασχόληση. Αυτή η δέσμη λοιπόν ή το πακέτο θα είναι το θεμέλιο της οικονομικής πολιτικής μας. και να βρούμε τα στοιχεία ε, βάσει των οποίων τα κράτη-μέλη θα συντονίσουν τις πολιτικές τους. Έτσι λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω παραμένει πάρα πολύ σημαντική και κρίσιμη εξή φάση. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φέρει την εξέταση, την ετήσια της ανάπτυξης, θα έχουμε διπλή διάσταση ως προς το ρόλο μας. Δηλαδή να εξετάσουμε με ποιο τρόπο τα κράτη-μέλη έχουν ε, ολοκληρώσει το προηγούμενο οικονομικό έτος, νη πλην ένα, και ε, πώς θα χαράξουμε τη στρατηγική για το επόμενο έτος, νη συν ένα. Αυτό χρειάζεται βέβαια επαλήθευση και έλεγχο, αλλά νομίζω ε, κάπως έτσι φαντάζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα κυλήσουν τα πράγματα. Για το επόμενο έτος στους μεγάλους προσανατολισμούς δίνει ε, την έγκρισή του το Εαρινό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν είναι ο χώρος για το συντονισμό. Από εκεί και πέρα είναι η μεταφορά στην πράξη από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, κύρωση ε, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο και μετά τα, ε, τα κράτη-μέλη θα έχουν καταθέσει τα σχέδια τα εθνικά σχέδια, εν πάση περιπτώσει, μεταρρυθμίσεων για ε, το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Αυτή η φάση λοιπόν του συντονισμού πριν το Ερνό Συνέδριο είναι, συμβούλιο, συγγνώμη, είναι κρίσιμη. Ε, όχι να οργανωθούμε και να πούμε τι θα κάνουμε, ψηφίσματα, πολιτικές ομάδες ή οι κοινοβουλευτικές επιτροπές. Όχι. Θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε ένα διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, επαληθεύσουμε, για να εξακριβώσουμε πώς μπορούμε ακριβώ να επηρεάσουμε τη διαδικασία αυτή. Και σε τούτη την Επιτροπή και στην Επιτροπή Επασχόλησης είχα κάνει μια πρόταση. να θεωρήσουμε σχεδόν ομοθετικά κείμενα ε, με τροπολογίε και ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και τους μεγάλους προσανατολισμούς και τη της οικονομικής Αυτό που είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε είχαμε συνάντηση ε, με τα Εθνικά Κοινοβούλια και να έχουμε αυτή τη συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια πριν το Εαρινό Συμβούλιο, ακριβώς για να συντονίζουμε την οικονομική πολιτική, όπως σας είπα, ίσως θα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία αυτή έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη επιρροή στο συντονισμό αυτών των πολιτικών. Στη δεύτερη φάση του έτους, το δεύτερο εξάμεινο, δηλαδή μετά το Ερεινό Συμβούλιο και τη στιγμή που τα κράτη-μέλη έχουν βάλει, ε, στο, έχουν δρομολογήσει ας πούμε κοινοτικά τα προγράμματα τους για τις μεταρρυθμίσεις, θέλουν να υπάρχει αυτή η λεγόμενη δημοσιονομική διάσκεψη. Δεν ξέρω να το σκεφτούμε αυτό για τον προπολογισμό, γιατί είναι άλλη μια ευκαιρία για συζήτηση. Και τέλος, αυτό που βλέπουμε να υπονοούν πολλές νομοθετικές εκθέσεις ε, ε, ε είναι το εξή. Ε, όταν ένα κράτο μέλο αντιμετωπίζει δυσκολίε, θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επεμβαίνει ω δημόσιο χώρο έκφραση, εξέταση τη κατάσταση των ιδιαίτερων δυσκολιών. Όταν ήρθε ο Γιώργος Παπανδρέου στην Επιτροπή της Κρίσης να παρουσιάσει την κατάσταση στη χώρα του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε θαυμάσια το ρόλο του. Ήταν εδώ στις Βρυξέλλες ένας χώρος δημόσιας συζήτησης. Όχι ε, καταγγελιών, όχι κατηγορίας, όχι κριτικής, αλλά χώρου δημόσιας έκφρασης. Αυτά λοιπόν για την έκθεση πρωτοβουλία την οποία μου αναθέσατε. Θα ήθελα να πω ότι από τεχνική πλευρά η ιδέα επί τη ουσία είναι να δούμε ποια θα είναι η εντολή ε, για να διαπραγματευτούμε μια διοργανική συμφωνία. Διότι η καλή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου εξαρτάται πολύ από τη δυνατότητα ελέγχου που έχουμε από την εμπειρογνωμοσύνη μας και όχι μόνο, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει κείμενα στα οποία να έχουμε και λόγο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λαμβάνει υπόψη του αυτά που θα έχουμε εμείς να πούμε κατά τη διάρκεια των επόμενων ε, οικονομικών ετών. Αυτά, Πρόεδρε, μπορεί να μακρηγόρησα, αλλά ε, ήθελα να σας εξηγήσω ακριβώς πώς βλέπω ε, αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ. Θα έχουμε χρόνο να το διερευνήσουμε αυτό και τις διάφορες επιλογές και κατευθύνσεις που θα θέλαμε να ακολουθήσουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα γι' αυτό. Μπεν Χάρτε, ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περβάνς ε, για αυτά τα οποία είπε και να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις για το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Ο Ζαν Πολ δεν είναι εδώ, μου ζήτησε όμως ε, να πω λίγα λόγια. Κατά την απόψή μου, πράγματι, όλοι εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο πρέπει να αγωνιστούμε έτσι ώστε ο ρόλος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων να ενισχυθεί σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να έχουμε μια εντονότερη ανταλλαγή απόψε με τους συναδέλφους στα εθνικά κοινοβούλια, οπότε χαιρετίζω αυτό το οποίο είπε η Περβάνς. Επίσης θεωρώ πως η πρόκληση θα είναι το πώς ε, στο μέλλον ε, θα μπορέσουμε να συντονίσουμε την οικονομική πολιτική. Δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για επιτήρηση για εμένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας. Κάτι το οποίο είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Γι' αυτό θεωρώ πως ε, για μένα προσωπικά και για την ομάδα μας ε, είναι αυτό ένα σημείο κλειδί όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπωσδήποτε έχουμε και κάποιες αμφιβολίες για τα ζητήματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουν, να συζητήσουμε για τη σχέση τελικά του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με όλο αυτό το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, και με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Αυτά είναι όλα ζητήματα τα οποία πρέπει να ανοίξουμε και να ξεκαθαρίσουμε τους τελευταίους μήνες. Συνελώνται Πρέπει να δούμε τον στόχο μας, τον τελικό, δηλαδή θέμε οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και αύξηση της απασχόλησης, οπότε θα πρέπει να δούμε τα μέτρα του ε, Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω δύο ακόμα ομιλητές, Βίκη και Ζουζέ. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Περβάνς ε, για τα σχόλιά της. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ στο δικό μου κράτος μέλος και σε άλλα κράτη-μέλη σε όλους τους πολιτικούς αλλά και κυρίως μεταξύ των πολιτών είναι μια επιθυμία να αντιληφθούμε από πού προέρχονται και πού πηγαίνουν τα δημόσια χρήματα και διαφάνεια και εμπιστοσύνη σε αυτό το σύστημα. Η διαφάνεια, η ανεξαρτησία των προβλέψεων, τα αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία είναι πράγματα τα οποία ζητάει το κοινό μετά από αυτά τα οποία είδε σε διάφορα κράτη-μέλη. Για εμένα ο ρόλος του εξαμήνου είναι κλειδί για να δοθεί αυτό το επίπεδο λογοδοσίας και διαφάνειας. Αλλά βεβαίως ε, είναι και τα ζητήματα που εξής η ποιοι είναι οι αριθμοί που θα μοιραζόμαστε, πόσο ε, στιβαρές είναι οι διαδικασίες πρόβλεψης, ε, τι πληροφορίες θα μπαίνουν σε αυτό το εξάμεινο και η ανεξαρτησία από τους πολιτικούς οποιασδήποτε απόχρωσης έτσι ώστε τα νούμερα αυτά να είναι αξιόπιστα για το κοινό μας. Η συνάντηση που είχαμε φέτος με τα Εθνικά Κοινοβούλια ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Είχαμε μια μισή ημέρα συνεδριάσεων και γνωρίζω πως η πρόεδρος μας ήταν μια μισή ημέρα στην Πρόεδρια. Ήταν πολλά και ενδιαφέροντα τα ερωτήματα από εθνικούς βουλευτές και ευρωβουλευτές και Νομίζω πως μπορούμε άρα να βασιστούμε σε αυτό και να έχουμε αυτή την ανοιχτή συζήτηση, αυτό το φόρουμ και μετά θα πρέπει να ζητήσουμε νομίζω μια ανοιχτή συζήτηση για να ε, συνεισφέρουμε κι εμείς και βεβαίως πρέπει να παίξουμε κι εμείς τον ρόλο μας ε, ε, στο διάλογο μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Uh, το άλλο ζήτημα που βλέπω από πολλά κράτη-μέλη και μέλη του κοινού είναι πως όταν βλέπουν αυτό το εξάμεινο λένε εντάξει καλή διαφάνεια αλλά πόση διαφάνεια υπάρχει όταν φτάνουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο και, και αυτό το χρωστάμε στο κοινό μας. Δηλαδή μπορούμε να συζητάμε για το μέγεθος ή το μη μέγεθος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού αλλά σε μας επαφίεται να δείξουμε πως υπάρχει εξίσου διαφάνεια και στο ευρωπαϊκό επίπεδο από πού προέρχονται και πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά και νομίζω πως πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Έχουμε πολλές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες εδώ πέρα για να δοθεί αυτή η διαφάνεια στο κοινό και η ανεξαρτησία που για μένα είναι θέμα κλειδί. Ευχαριστώ. Έχουμε και άλλους ομιλητές τώρα, τον Λίαμ και τον Σβέντζοζε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Μπερές που μας παρουσίασε την εργασία της, γιατί αυτό μου επιτρέπει να προβώ σε κάποια σχόλια. Και τα σχόλια αυτά τα κάνω για να προσπαθήσω να βελτιώσω αυτό που έχουμε επιτάπητο. Δηλαδή, ποια είναι η προστιθέμενη αξία που εμείς μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτό το πακέτο σε Ευρωκοινοβούλιο. Και θα κάνω κάποια σχόλια προσπαθώντας να είμαι κάπως ε, οργανωμένος. Καταρχήν, το Συμβούλιο των Υπουργών έχει αναλάβει αυτή, έχει μάλλον υιοθετήσει αυτή την ιδέα. Είναι μια μορφή νομοθεσία, ένα πρότυπο νομοθεσία όπου οι Υπουργοί Οικονομία και Οικονομικών παίζουν σημαντικό ρόλο. Φυσικά το Κοινοβούλιο μπορεί και αυτό να παρέμβει, αλλά όχι αρκετά κατά τη γνώμη μου για αυτό το Ευρωπαϊκό Εξάμενο. Για να αποφευθεί λοιπόν ένα τέτοιο πρόβλημα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατευθύνουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο όσον αφορά την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και το γενικότερο πακέτο που έχουμε ξεκινήσει για να αποφύγουμε την επανάληψη μιας κρίσης. Δεύτερο σχόλιο. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο από πολλές απόψεις δεν είναι συνεπές με τα υπόλοιπα μέτρα για τα οποία μίλησε πριν από λίγο. Ξέρω πως έχουμε μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό. Υπάρχουν ε, οι οικονομικές ανισορροπίες και το σύμφωνο Ευρώ μια ολόκληρη σειρά λοιπόν πραγμάτων που βρίσκουμε στο πακέτο αυτό. Δεύτερο πρόβλημα είναι πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη επίσης τους μηχανισμούς διάσωσης. Μηχανισμοί διάσωσης προσωρινοί όπου γνωρίζουμε ότι δεν έχουν λειτουργήσει καλά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χρειάστηκε να μειώσει τις συνθήκες για την Ελλάδα, για την Ιρλανδία είναι έτοιμο να το κάνει, με την προπόθεση ότι η Ιρλανδία θα κάνει μια προσπάθεια όσον αφορά την δημοσιονομική ε, πειθαρχία. Άρα λοιπόν αυτός ο οριστικός μηχανισμός διάσωσης, κατά τη γνώμη μου, ε, περιέχει τα ίδια μειονεκτήματα όπως ο προσωρινός μηχανισμός και προσθέτει και κάποια επιπλέον μειονεκτήματα, γιατί καταρχήν υπήρξαν οι δηλώσεις της κυρίας Μέρουκελ που είπε ότι πρέπει να υπάρχει και ιδιωτική συμμετοχή, πράγμα που προκάλεσε την πτώση της Ιρλανδίας, σχόλια της ε, ΕΚΤ, που οπότε μια τέτοια δήλωση αυξάνει την πτυτικότητα των αγορών, πράγμα που έγινε και όλα στην πράξη. Ο καθένα δίνει τη δική του απόχρωση, λέει ότι θα γίνουν τα πράγματα αναπερίπτωση, αυτό όμω δεν προσφέρει τίποτα. Έπειτα λέμε ότι θα ισχύουν όλα αυτά από το 2013, πράγμα το οποίο είναι αντιφατικό και μας λένε επίσης ότι θα σεβαστούν τα όσα λέει το Δουνουτού. Δηλαδή και άλλο λάδι στη φωτιά στην ουσία. 2013 Άρα λοιπόν ο ιδιωτικό τομέα δεν θα συμμετέχει στην αναδιάρθρωση του χρέου μέχρι το 2013. Από το 2013 και μετά, ναι. Αν από το 2013 και μετά δηλώσουμε ότι δεν είναι πλέον βιώσιμη η οικονομία μια χώρα, αυτό θα έχει επιπτώσει και στα αξιόγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από αυτή την ημερομηνία. Άμα μια χώρα δεν μπορεί να πληρώσει το νέο χρέο, δεν μπορεί να πληρώσει ούτε και το παλιό. Και είναι πολύ σημαντικό έπειτα αυτό που λέει για το Δουνουτού. Ότι δηλαδή μόνο μία περίπτωση υπήρξε όπου το Δουνουτού ε, ανέτρεξε στην αναδιάρθρωση του χρέους ήταν το 2003 στην Αργεντινή. Ε, απευθύνθηκαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέγοντας ότι ναι, ναι θα το αποπληρώσουμε. Η έκπτωση ε, παραμένει πάντα και υπάρχει πάντα και ένας μηχανισμός που επιτρέπει στην Αργεντινή να αξιολογήσει τι κάνουν άλλες χώρες που βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Τώρα, ποιο άλλο μειονέκτημα έχει αυτός ο μηχανισμός οριστική, οριστική τελικός μηχανισμός διάσωση. Δεν είναι απόλυτα αντικειμενικό για τη γνώμη μου και αυτό είναι το χειρότερο για την αγορά. Γιατί η αγορά ε, χρειάζεται σταθερότητα και βεβαιότητα. Συμπέρασμα. Κατά την άποψή μου, αυτό που χρειάζεται είναι το εξή. Οι πολιτικέ απαντήσει των κυβερνήσεων στι συστάσει που γίνονται για το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα πρέπει επίση να λαμβάνονται υπόψη τη στιγμή ε, που ε, έρχεται η ώρα τη απόφαση αναδιάρθρωση ή όχι του χρέου αν γίνει αυτό θα πάμε και σε ένα ε, σωστό μηχανισμό. Και τελειώνω. Υπάρχει μια ακόμα ιδέα της Προέδρου που λέει ότι θα πρέπει να συνδέσουμε το μηχανισμό διάσωσης, την αναδιάρθρωση του χρέους με το σύστημα ε, ε, κρίσης και κανονισμού της κρίσης των, κρατών, των τραπεζών. Σήμερα ισχύει το θεώρημα ότι τα κράτη δεν χρεοκοπούν. Ε, θα πρέπει όμως να υπάρξει ένα σύστημα υπολογισμού των συντελεστών κεφαλαίου. Ένα ε, συνολικό μοντέλο χρειάζεται, το οποίο ακόμα δεν έχουμε ορίσει, δεν έχουμε σωματώσει, δεν έχουμε διευκρινίσει, γι' αυτό έχουμε ανεπάρκειες ή επικαλύψεις και αυτό που χρειάζεται το Κοινοβούλιο να κάνει ακριβω αυτό. Να δει ποιο είναι το τελικό σχέδιο, η τελική εικόνα, πού θέλουμε να πάμε και να συμπεριλάβουμε όλα αυτά ε, στα διάφορα εγχειρήματά μας. Ο μηχανισμός είναι ακόμα εκτός και ο προσωρινός και ο μόνιμος, η επίλυση της τραπεζικής ε, κρίσης. Και ε, ένας Ισπανός ποιητής έχει πει ότι δεν υπάρχει ποτέ ούριος άνεμος όταν δεν ξέρεις πού πηγαίνει στη θάλασσα. Συμφωνώ. Μετά όσα είπατε, ότι το χρέος είναι το μεγάλο ε, ζήτημα. Είναι σαν ένας ελέφαντας να ήταν εδώ μέσα στην αίθουσα. Δεν μπορούμε να κάνουμε το αγνοούμε για να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Ο Λέω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περβάονς που επέμεινε για ένα σημαντικό θέμα που είναι ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών και επί του οποίου στην ουσία επικρατεί η εποπτεία. Γιατί διάβασα την οδηγία, διάβασα τις τροπολογίες που πρότειναν διάφοροι συνάδελφοι στο πλαίσιο του πακέτου για τη διακυβέρνηση και έχω την αίσθηση ότι το περιοριζόμαστε και δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για συντονισμό σε θέματα μακροοικονομικής πολιτικής. Η αίσθηση που δίνει η ανάγνωση της οδηγίας και των τροπολογιών είναι ότι ε, ενισχύουμε και καθιερώνουμε τον προκυκλικό χαρακτήρα των οικονομικών πολιτικών που έχουν εγκατασταθεί στην Ευρώπη εδώ και κάποιο καιρό. Και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι απαγορεύουμε από εδώ και μπρο τη δυνατότητα αντίδραση με βάση τη συγκυρία. Ανάλογα μάλλον με τη συγκυρία. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί οι συγκυρίες σε διάφορε χώρε δεν είναι οι ίδιες και πιο συγκεκριμένα η ευρωπαϊκή η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι κατάλληλη για πολιτικές ε, ε, δημοσιονομικής ε, παγίες. Αν δούμε το αποσοστά ε, παραγωγικής δυνατότητας. Πιστεύω ότι είμαστε 6 με 8% κάτω από τη χρήση των παραγωγικών δυνατοτήτων μας. Αυτό σημαίνει πως μια αυξημένη υποπτία των δημοσιονομικών πολιτικών που θα θέλαμε ε, να είναι πολύ αυστηρές και λιτές, δηλαδή πολιτική λιτότητας, θα είχε αυτό πολύ αρνητικές επιπτώσεις σε αυτή την περίοδο και δεν θα κατάφερνε να μειώσει και τα ελλείμματα. Τώρα, όσον ε, σε σχέση με όσο είπε ο κύριος Γκαρσία Μαργκάριου. Εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να βάλουμε επιτάπητο στο ευρωπαϊκό εξάμεινο την αναδιάρθρωση του χρέους. Γιατί όταν δούμε το αίτια της αύξησης του χρέους και εδώ πρέπει να δούμε κάτω από το επίπεδο της θάλασσας για να δούμε το παγόβουνο ολόκληρο, θα διαπιστώσουμε ότι δεν έχουν κραγεί οι δαπάνε, αλλά οι, ε, τα έσοδα έχουν μειωθεί σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε, γιατί οι ευρωπαϊκέ χώρε άρχισαν ε, ε, πολιτικέ φορολογίες που στην ουσία αύξησαν το έλλειμμα. Αν δούμε, πούμε, την ελληνική περίπτωση, η κυβέρνηση Παπαδρέου κληρονόμησε μια κατάσταση για την οποία δεν είναι υπεύθυνη, όπου και άλλε κυβερνήσει έκαναν σφάλματα, αλλά το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους είναι ε, ένα θέμα απόλυτα κέριο. Και έπειτα για τις οικονομικές πολιτικές δεν είναι μόνο ο συντονισμός των πολιτικών ανάμεσα στα κράτη-μέλη, είναι και αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά το policy mix, δηλαδή ο συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών και των νομισματικών πολιτικών. Και ως προς αυτό η Περβαός έθιξε ένα πρόβλημα κλειδί που είναι το πρόβλημα της σχέσης ανάμεσα στην δημοσιονομική πολιτική των κρατών μελών και της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Και εδώ λοιπόν που λέω ο νομισματικός διάλογος με την ΕΚΤ έχει μετατραπεί σε διάλογο κοφών. Για παράδειγμα, τα επιτόκια αυτή τη στιγμή που είναι σήμερα το μόνο μέσο δράσης για την μακροοικονομική συγκυρία ε, ε, ε, συνδέονται, μάλλον χρησιμοποιούνται με περιοριστικό τρόπο. Και ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας μας το ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα στον τελευταίο νομισματικό διάλογο ότι θα σκληρύνει η νομισματική πολιτική. Αυτό φαίνεται να είναι άτοπο σε αυτή την σημερινή κατάσταση. Και ένα σωστό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών θα έλεγε τουλάχιστον να το συζητήσουμε. Δεύτερη παρατήρηση πάντα για το χρέος, Του θέσαμε το ερώτημα κατά πόσο υπάρχει σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσα στην ε, αγορά του ελληνικού χρέους στη δευτερεύουσα αγορά και την αύξηση των επιτοκίων στο 15% ε, για τα ελληνικά δάνεια και δεν μας απάντησε δεν μας είπε τι θα κάνει με την αναδιάρθρωση του χρέους και πώς θα γίνει να έχουμε ένα καλό policy mix στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω πως η έκθεση της Περβάος Περές είναι μια καλή ευκαιρία για να θίξουμε όλα τα ταμπού στην Ευρωπαϊκή Κλίμακα. Ε, το Κοινοβούλιο δεν, ε, δεν φοβάται να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Νομίζω πως πρωτοπορεί. Ο Σβέν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις. Το ένα είναι, εάν δούμε τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη παρουσιαστεί, έχουν κυμαίνονται ως προς την ποιότητα και πρέπει να τα δούμε προσεκτικά γιατί κάποια από αυτά δεν ανταποκρίνονται στις ε, προκλήσεις και είναι ενισχυτικό. Αν δεν πάρουμε σοβαρά αυτή τη διαδικασία, ανεξαρτήτως του τι θα κάνουμε, δεν θα λειτουργήσει. Δεύτερον, συμφωνήσαμε σε πέντε στόχους ε, κλειδιά και πάρα πολλές πρωτοβουλίες ε, και θα πρέπει να μην περιοριστούμε μόνο σε μια στρατηγική ανάπτυξη, αλλά να είναι τόσο γενικό όσο και οι στόχοι που έχουμε. Και πρέπει να δούμε πόσους στόχους μπορούμε να ακολουθήσουμε, αλλά πρέπει να έχουμε ε, και το παραγωγικό δυναμικό. Αλλά βεβαίω αν δεν έχει μείνει πλανήτης, ε, δεν ωφελεί αυτό κανέναν. Δεν ξέρω αν ε, λοιπόν μπορούμε να κρίνουμε το, το μείγμα της πολιτικής. Ο Λίαν ξέρει σε τι αναφέρομαι. Επίσης υπήρχε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τηλεφωνική διάσκεψη μεταξύ μελών της Επιτροπής και της Γερμανικής Βουλής. Ίσως για να έχουμε υψηλότερο επίπεδο συμμετοχή από τα Εθνικά Κοινοβούλια θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια μέσα όπως η βίντεο διάσκεψη για να επιτρέψουμε και πραγματική συμμετοχή των αρμοδίων στις εθνικές επιτροπές. Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Εμείς λέμε πως είχαμε μια καλή συνεδρίαση αλλά δεν υπήρχαν αρκετοί ευρωβουλευτές. Συμφωνώ και εγώ και εμένα απασχολεί αυτό, έχετε δίκιο. Το θέμα είναι πως απ' την άλλη, εάν δείτε τη συμμετοχή των εθνικών ε, κοινοβουλίων, ήταν η συνήθις ύποπτη. Αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο για τα ευρωπαϊκά. Α, δεν μας βοηθάει να έχουμε δεσμευτικά αποτελέσματα. Πρέπει και αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν στα εθνικά κοινοβούλια να εμπλακούν. Οπότε θα πρέπει να βρούμε μια διαδικασία για να έχουμε κάποια σχέση με τους εθνικούς βουλευτές, γιατί υπάρχει ένας υπόγειος ανταγωνισμός, όχι μόνο μεταξύ των κυβερνήσεων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και στα εθνικά κοινοβούλια ανησυχούν για εμάς. Οπότε, για να το αποφύγουμε, πρέπει να έχουμε μια συνεργασία. Τέλος, στην όλη αυτή διαδικασία του εξαμήνου, πρέπει να φροντίσουμε να μιλήσουν και οι κοινωνικοί εταίροι και να αποτελέσει αυτό το τμήμα της ε, όλης ε, διαδικασίας. Μα αναμένω λοιπόν να, εργαστεί η από αυτού. Καλή οικονομική ανάπτυξη, αλλά στο, στα όρια της ε, κοινωνικής ισότητας και τα όρια του πλανήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να σας πω πως ε, το Κοινοβούλιο ήδη είχε κάνει κάποιες, ε, κάποια βήματα για βιντεοδιασκέψεις. Το είδαμε στη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Ο κύριος Χουντής ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων δεν μπορούσα να είμαι εγκαίρος στη συνεδρίαση, στην έναρξη και να ακούσω και την εισηγήτριά μας την κυρία Μπερές ε, ελπίζω ότι και ξέρω είμαι σίγουρος ότι θα ανέπτυξε ε, ενδιαφέρουσες σκέψεις. Ε, η πρώτη, ανάγνωση, η πρώτη συζήτηση μας επιτρέπει λοιπόν να ανταλλάξουμε ορισμένες σκέψεις. Πρώτον, αύριο μεθαύριο ο Έλληνας Πρωθυπουργό θα εξαγγείλει στο Υπουργικό Συμβούλιο και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και κατά συνέπεια στον ελληνικό λαό ένα νέο πακέτο μέτρων ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να μπορέσει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ελλείμματος και του χρέους. Αυτά τα μέτρα θα είναι σκληρά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Σημαίνουν περαιτέρω μείωση των μισθών, περαιτέρω μείωση επιδομάτων, σκληρά αντικοινωνικά μέτρα. Μία από τις αιτίες εξαγγελίας αυτών των μέτρων είναι ότι έπεσαν έξω οι προβλέψεις για πιθανά έσοδα που θα ανακούφισαν κάπως την κατάσταση. Και αναδεικνύεται το πρόβλημα που ανέφερε και ο συνάδελφος πριν, ότι και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες το πρόβλημα που σήμερα εμφανίζεται ότι είναι ανεξέλεκτο, δηλαδή <clears throat> το δημόσιο χρέος δεν είναι πρόβλημα δαπανών, αλλά κυρίως είναι πρόβλημα εσόδων. Κυρίως είναι πρόβλημα εσόδων. Γιατί είναι πρόβλημα εσόδων. Διότι εδώ και πολλά χρόνια η φορολογική πολιτική που ακολουθούνταν ήταν γεμάτο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, <clears throat> απεριόριστες φοροαπαλλαγές, υπήρχε μεγάλη φοροδιαφυγή και βεβαίως υπήρχαν και ζητήματα δαπανών και επιτρέψτε μου να σας πω, ε, είμαστε από τον πολιτικό φορέα, ο μόνος πολιτικός φορέας στην Ελλάδα που επιμέναμε ότι δεν έπρεπε η Ελλάδα με την οικονομική δυνατότητα που είχε να αναλάβει τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων όπου έγινε μεγάλη δαπάνη και δεν νομίζω ότι μας άφησε και τίποτα πέρα από τη δόξα. Αν υπάρχει και αυτή. Λοιπόν, σήμερα αυτό το πρόβλημα δεν φαίνεται να έχει άκρη. Και δυστυχώς αποδεικνύεται ότι η επικέντρωση στο πρόβλημα του δημοσίου χρέους και μάλιστα ως αιτία της κρίσης μας οδηγεί σε λάθος ατραπούς, σε λάθος δρόμους. Κατόπιν τούτου τα μέτρα που συζητούνται όπω στην προκειμένη περίπτωση, αν δεν κάνω λάθο, συζητούμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο, είναι πολύ συζητήσιμη και αμφίβολη αναποτελεσματικότητα. Κατ' εμέ, σε σχέση με το ευρωπαϊκό εξάμεινο και τον προέλεγχο των εθνικών προπολογισμών, εγείρει θέμα συνταγματική και δημοκρατική τάξη. Αν από τα εθνικά κοινοβούλια αφαιρεθεί μία από τι βασικέ αρμοδιότητε να ψηφίζουν όπως ψηφίζουν τον προϋπολογισμό και αυτό ενταχθεί μέσα σε έναν προέλεγχο σημαίνει ότι πολιτικά δεν υπάρχει δυνατότητα να ασκήσεις εναλλακτικές πολιτικές. Αυτή η αναφορά αγαπητοί συνάδελφοι μου θυμίζει την απέτηση του νέου συμφώνου για το Europlus που εκτός των άλλων θέλει όλες αυτές τις δεσμεύσεις να περάσουν είτε στο Σύνταγμα είτε να πάρουν ένα νομικό δεσμευτικά χαρακτήρα και κατά τη γνώμη μου είναι πρόβλημα δημοκρατίας και πρόβλημα νομιμοποίησης πέρα από το ότι δεν συγκροτεί κατά την άποψή μας και κατά την άποψή μου ξεπέρασμα της οικονομικής ε, κατάστασης, ε, των προβλημάτων. Τελειώνω. Ναι, συντονισμός των οικονομικών πολιτικών. Αλλά με, με δύο-τρεις προϋποθέσεις τις αναφέρω γρήγορα για να μην φάω το χρόνο. Πρώτον, πρέπει να αναγνωριστεί ότι το πρόβλημα του χρέου είναι πανευρωπαϊκό και όχι μόνο των τριών χωρών που σήμερα είναι είτε στο μηχανισμό είτε θα μπουν. Και ενώ την Πορτογαλία. Είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα και επομένω πρέπει να βρεθούν τρόποι πανευρωπαϊκής αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Δεύτερο, η αιμονή στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα είναι αντι η αναπτυξιακή, αντικοινωνική θα βυθίσει στην ύφεση. Η ύφεση όπως ξέρετε στην Ελλάδα που ήδη είναι πάνω από τις προβλέψεις είναι μείον 6. Στο τελευταίο τρίμηνο τουλάχιστον του προηγούμενου χρόνου ήταν μείον 6 ύφεση. Τι έσοδα να έχει με τέτοια ύφεση, με τέτοια ανάπτυξη εντό εισαγωγικών ανάπτυξη. Πού θα τα βρει τα έσοδα, πώ θα λύσει το πρόβλημα. Μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο. Επομένω, δεύτερο, να αλλάξει το σύμφωνο σταθερότητα. Και το τρίτο, και το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης πολύ φοβούμαι ότι είναι ένα μοχλός πίεσης για μεγαλύτερες περικοπές, για περισσότερες αλλαγές και σήμερα στην πρώτη γραμμή και τελειώνω με αυτό που ξεκίνησα η απέτηση είναι να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές. Είναι αυτό που απαιτεί εν τέλει το δεύτερο σκέλος της οικονομικής διακυβέρνησης, δηλαδή η επιτήρηση των μακροοικονομικών ισορροπιών. Επειδή η επιτήρηση σημαίνει και κάποιους δείκτες που δεν εξαρτώνται από το κράτος, εξαγωγές και τα λοιπά και άλλα τέτοια πράγματα, σημαίνει ότι θα πάμε σε συνεχείς αναδιαθρώσεις. Αυτές είναι οι σκέψεις μας. Έχω τη γνώμη ότι όλο το πακέτο και η λογική κινείται σε λάθος κατεύθυνση και δεν θα μας βγάλει από τα προβλήματα, δεν εννοώ της Ελλάδας πια γιατί δεν είναι το πρόβλημα μόνο ελληνικό, αλλά θα μας βγάλει έξω από μια λογική μιας Ευρώπης που αντιμετωπίζει την κρίση θα προσέθετα και την τελευταία λέξη γιατί έχει ξεχαστεί με μια αίσθηση αλληλεγγύης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω πως αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Οι χώρες που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα οι πυροσβέστες αν θέλετε γίνονται ειδικοί γιατί αντιμετωπίζουν το, το ζήτημα εκ του συνεγγύς και είναι σιωπηλοί και δεν μιλούν λόγω των διεθνών αγορών και τα λοιπά. Και αυτούς πρέπει να ακούσουμε. Άντε αυτού ακούμε τους άλλους που είναι άμομοι, αν θέλετε, και λένε ηθικολογίες. Τις ε, προάλλες ε, διάβαζα τον Σμάργκη από κάποια κεντρική τράπεζα που έλεγε πως φορολογούμενοι έτσι τους αξίζει να υποφέρουν γιατί αυτοί όρισαν τις ρυθμιστικές αρχές που είχαν ε, την τάδε ρύθμιση που άφηνε ε, την ε, γάτα, τα ποντίκια να χορεύουν σε ολυμπικά κτλ. Δηλαδή είναι ο χειρότερος συντηρητισμός των τραπεζικών και δεν βοηθάει να βρεθεί μια λύση. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες που λένε να είμαστε ευέλικτοι. Δεν είναι θέμα ευελιξίες. Πρέπει να έχουμε περισσότερες διεξόδους. Ξέρετε πως οι διέξοδοι, οι παλαιοί οι παλαιές έχουν ε, κλείσει της υποτίμησης ε, συμπεριλαμβανομένης. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτό το πακέτο διακυβέρνησης και να είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα. Και ε, δεν βλέπω πως αυτό μόνο του θα μας βγάλει από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ευχαριστώ. Θα κάνω και εγώ κάποια σχόλια μετά από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Χούντης για το ότι στο εξάμεινο αυτό αφαιρούμε τις ε, εξουσίες των Εθνικών Κοινοβουλίων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τα Εθνικά Κοινοβούλια, εδώ πέρα, Κάποια από αυτά σχολίασαν πως ε, συμβαίνει το αντίστροφο. Για πρώτη φορά ένιωθαν μέρος της ε, διαδικασίας ε, στο επίπεδο της Ένωσης. Και αυτή είναι η γραμμή που θα πρέπει να ενισχύσουμε νομίζω για να θεωρήσουν και στο εθνικό επίπεδο πως είναι δική τους υπόθεση αυτό το πράγμα. Αυτό νομίζω χρειάζεται να πω γιατί συμφωνώ με πάρα πολλά από αυτά τα οποία ακούστηκαν ως το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης, αν και περιέχει πολλά θετικά πράγματα για να μας βγάλει από το πρόβλημα, ακόμα δεν επαρκούν τα μέτρα, ειδικά για τις ε, χώρες εκείνες οι οποίες είναι σε δυσκολία. Και δεν θα καταφέρουμε να επανέλθουν σε μια βιώσιμη πορεία εάν ε, μόνο τις κάνουμε να πληρώνουν πολύ περισσότερο και αντλούμε προσόδους. Περβάνς, θα ήθελες να σου πει κάτι η Κομισιόν? Αν έχει κάτι η Κομισιόν, ας μας πει τι γίνεται με το τρέχον εξάμεινο και μετά έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κάποια σύντομα σχόλια. Πρέπει να δούμε τη φύση του ευρωπαϊκού εξαμήνου δεν αφορά μόνο την επιτήρηση, είναι θέμα συντονισμού με βάση κάποιες ε, καθορισμένες ε, προτεραιότητες, ε, με βάση την Ευρώπη 2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Οπότε βασίζεται σε μία προσέγγιση συντονισμένη για τη μακροοικονομική πολιτική, όπως εκφράζεται μέσω αυτών των κατευθυντήριων γραμμών. Πρέπει να τονίσουμε πως η επιτήρηση βεβαίως δεν είναι ε, ένα σκληρό μέσο, είναι ένα ήπιο μέσο. Μπορεί όμως να βελτιωθεί και, στο, και αυτό μπορεί να γίνει, θεωρεί η Κομισιόν, με δύο τρόπους. Πρώτα απ' όλα να έχουμε μια συνολική προσέγγιση όσον αφορά αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής και απασχόλησης και το να δούμε συνεκτικά το φάσμα των οικονομικών πολιτικών δίνοντας εξίσου βάρος στους στόχους που έχουν τεθεί. Και τρίτον, να τονίσουμε βεβαίως πως πέρα από το ευρωπαϊκό εξάμεινο και πέρα από την επιτήρηση υπάρχουν και μηχανισμοί επιβολής. Δεν σταματάει δηλαδή η υπόθεση με μία έκθεση της Κομισιόν ή του Συμβουλίου για τα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα. Συνεχίζεται με συστάσεις που υιοθετεί το Συμβούλιο και αξιολόγηση συμμόρφωσης με αυτές τις συστάσεις. Αυτό λαμβάνει χώρα βεβαίως εκτός του πλαισίου του εξαμήνου, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να αποτελέσει ένα τρόπο να διασφαλίσουμε πως υπάρχει συντονισμός, αυξημένη επιτήρηση και επιβολή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου όσον αφορά την Ένωση, την Ευρωζώνη και σε κάποιες περιπτώσεις ε, και με μονομένα Το δεύτερο σημαντικό πράγμα που πρέπει να πούμε είναι πως το ευρωπαϊκό εξάμεινο πρέπει να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Είναι ένα μέσο με στόχο να βγούμε από αυτή την κρίση και να βελτιώσουμε την ε, προσέγγιση μας για την οικονομική πολιτική στο μέλλον. Και άρα, σωστό είναι να δούμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο ένα μέσο μεταξύ άλλων που έχει προτείνει η Κομισιόν ως απάντηση στην κρίση. Και τέλος να τονίσω πως η Κομισιόν βεβαίως εξακολουθεί να θέλει την ε, συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια και την ε, εισηγήτρια για να ορίσουμε με τρόπο σύμφωνο προς τη συνθήκη τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο ίδιος ο Επίτροπος και ο Πρόεδρος της Κομισιόν ε, έχουν επαναλάβει πολλές φορές την δέσμευσή μας για να βρεθεί ο σωστός ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και σε ό,τι συνδέεται με αυτό. Και βεβαίως ε, θα συνεργαστούμε στενά με την εισηγητριά σας για να πετύχουμε αυτό ακριβώς. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάω. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δίκιο είχατε που δώσατε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεισέφερε πάρα πολύ. Επιβεβαίωσε τι σημαίνει lip service. Ε, τα λόγια. Ε, τα λόγια. Θα πρέπει να ε, προσέξουμε πολύ το ρόλο του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για τη συνεισφορά αυτή και χάρη στην έκθεσή μου ελπίζω να ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο, αυτή την κατάσταση της συνειδητοποίηση του δημοκρατικού διακυβεύματος γύρω από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Συγγνώμη, αλλά όταν γυρνάω στη χώρα μου, ο κόσμος συζητάει λίγο, καταλαβαίνει τι τρέχει ότι οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών θα καθορίζονται απολύτως και πάρα πολύ αυστηρά εκτός του δημοκρατικού διαλόγου. Μα τι απομένει για το εθνικό δημοκρατικό ε, γίγνεσθε. Το θέμα της δημοκρατίας δεν είναι ότι Α, για να δούμε τι ρόλο θα καθίσουμε να σκεφτούμε να επινοήσουμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έκλεισε το μικρόφωνο. Ε, Κανονικά δουλεύει. Εντάξει, επίσημα τουλάχιστον αυτό λέει εδώ ανάβει. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για τα όσα είπανε. Ε, κατανοώ ε, ορισμένες τοποθετήσεις βεβαίως απορρέουν από το περιεχόμενο της πολιτικής και τι θα... Ε, ασκηθεί περισσότερο από την έκθεση πρωτοβουλίας που είναι έκθεση διαδικαστική και εγώ μιλώ για τη ε, λειτουργία της δημοκρατίας. Αυτό με ενδιαφέρει. Έχει ε, κάποια χρησιμότητα λοιπόν και προς τα εκεί. Ε, σε σχέση με τα εισαγωγικά σχόλια θέλω να κάνω δύο συμπληρωματικές παρατηρήσεις που δεν είχα ευκαιρία να πω προηγουμένως, δεν είχα το χρόνο, αλλά είναι σημαντικές για τη συζήτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέθεσε μια μελέτη σε ένα εξωτερικό συνεργάτη, σε ένα Ινστιτούτο, για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και να έχουμε ζήτημα αξιολόγησης, εκτίμησης. Αυτό που είπε ο Σβέν Γκίγκολτ, πούμε, αυτά που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, βάση εργασίας θα πρέπει κάπως να τα ε, έχουμε υπόψη μας. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να δούμε πώς η δημοσιονομική συζήτηση διεξάγεται στα κράτη ε, που είναι ομοσπονδιακά ή συνομοσπονδιακά. Ένα από τα θέματα που μας απασχολεί εδώ είναι και αυτό. Δηλαδή, όταν σε ένα κράτος υπάρχουν κυρίαρχες οντότητες ε, που διαχειρίζονται το δικό τους προϋπολογισμό ε, στη συνέχεια καλείστε αυτά να τα συγκεντρώσετε σε ένα συνολικότερο επίπεδο. Επίσης και το θέμα των ε, προθεσμιών. Πριν εφεύρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη νέα ιδέα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, είχαμε αυτή τη δυσκολία έτσι κι αλλιώς. Τότε τι είχαμε, τις μεγάλες ε, πολιτικές και οικονομικές κατευθύνσεις και τις κατευθύνες γραμμές για την απασχόληση. Και από τότε σπαζοκεφαλιάζαμε για να βρούμε ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να επέμβουμε, για να αναγκάσουμε το Συμβούλιο να λάβει υπόψη του αυτά που έχουμε να πούμε. Και τώρα χειροτερεύουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα, διότι αν θέλουμε να λειτουργεί η δημοκρατία, τα εθνικά σχέδια μεταρρυθμίσεων, για παράδειγμα, θα πρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να μπορούν να τα εξετάζουν πριν τα διαβιβάσουν οι κυβερνήσεις στις Βρυξέλλες, εάν θέλουμε να υπάρχει αυτή η δημοκρατική λειτουργία. Ε, όμως, οι κυβερνήσεις επίσημα δεν μπορούν να συντάξουν τα εθνικά ε, σχέδια αυτά παρά μόνο μετά το Ερηνό Συμβούλιο και στη συνέχεια να τα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, τον Ιούλιο το καλοκαίρι, εν πάση περιπτώσει, να δώσει την ευλογία του το ε, Συμβούλιο. Να σα δώσω το χρονοδιάγραμμα για φέτος. Φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικυρώσει τις συστάσεις αναχώρα στι 7 Ιουνίου και στο Συμβούλιο θα πάει στη ΕΠΣΚΟ 17 Ιουνίου, 21 στο ΕΚΟΦΗΝ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 24 Ιουνίου. Εκεί μέσα πού παίζουν τα εθνικά κοινοβούλια. Και εμεί ε, που θα επέβουμε. και θεμα προθεσμιων κινητοποίηση ε καταλληλης χρονικης στιγμης και θα πρεπει εμεί να στοχευσουμε παρα λεπτό για να λέμε ε, τη γνώμη μας επιπατός εμπιστητού, γιατί θα τα κάνουμε όλα άσχημα και δεν θα επηρεάσουμε τίποτα. Πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. σε σχέση με τα όσα είπε η Βίκη Φόρτ που έφυγε, ε, τα πει κάποιο που θα τα ακούσει, για την ανεξαρτησία των στατιστικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν ανεξάρτητες και ποιοτικέ στατιστικέ. Αλλά δεν μπορεί η στατιστική να κάνει πολιτική αφενός και αφετέρου. Δηλαδή, λυπάμαι που έφυγε όμω. Πώ να το πω. είναι κάτι που με ανησυχεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν βλέπω να το συζητάμε με έντονο τρόπο. Δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά συνεχίζω να το λέω. Και σε σχέση με το όσο είπε ο Γκίγκολτ, αν θεωρούμε ότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν είναι κάτι αφηρημένο, αλλά είναι ένα στοιχείο σε μια ιεραρχία, σε ένα σύνολο, θα πρέπει να το οργανώσουμε αυτό το σύνολο. Και ο ακρογωνιαίος λήθος αυτής της συνεκτικής κατασκευής κανονικά είναι το 2020. Αυτό δεν είναι το βασικό δομικό στοιχείο, ο λήθος. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020 δεν μπορεί να πετύχει με τον ισχυρό προπολογισμό που έχει. Το έχουμε ξαναδεί, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όταν λοιπόν τα κράτη-μέλη καταθέτουν τους προπολογισμού τους, δίνουν τα δημοσιονομικά του στοιχεία, μα βοηθούν να κοιτάξουμε πώς ο δικός τους προϋπολογισμός συνεισφέρει και αυτός στην υλοποίηση του στρατηγικού στόχου μας για το 2020. Μα δεν είναι περίπλοκα αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ περίπλοκα, αλλά δεν το κάνουμε, δεν προχωρούμε και δεν είδα ακόμα στην έκθεση Vicky Ford ε, σημαντικά θέματα προς την κατεύθυνση αυτή. Ακούμε ότι το βασικότερο είναι η παιδεία. Συγγνώμη που βγαίνω από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αλλά προσπαθώ να πείσω ότι στην έκθεση της κυρίας Βίκη Φόρτ πρέπει να αναγκάσουμε τα κράτη-μέλη να καταθέτουν αυτό που στον προπολογισμό του συνεισφέρει στη στρατηγική για το 2020 της Ευρώπης. Σε σχέση με το όσα είπε ο συνάδελφος Γκαρσία Μαργκάγιο αναφέρθηκε στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και τους μεγάλους προσανατολισμούς για την οικονομική πολιτική. Εγώ αγωνίζομαι εδώ και καιρό για να συντονιστούν αυτά τα εργαλεία και τα μέσα, αλλά σας διαβεβαιώ ότι έχουν πεθάνει. Και πώς αποδεικνύεται αυτό. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτος ενέκρινε την ετήσια ανάλυση και έλεγχο της ανάπτυξης οικονομίας όπου προτείνει περικοπές μισθών και άλλα ενδιαφέροντα τεινά, δεν θεώρησε σκόπιμο και χρήσιμο να διορθώσει τους μεγάλους οικονομικούς ε, ε, προσαντολισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Είπε ότι είναι, ότι είναι συμβατά. Δηλαδή είναι μια άσκηση γραφειοκρατική, τυπική, ε, που δεν κοιτάει κάθε χρόνο ξεχωριστά τι γίνεται. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να έχει λόγο εκεί επίσημο, αλλά να προσαρμοστούμε σε αυτό που κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια ανάλυση και έλεγχο και όχι πλέον στις μεγάλες κατευθυντήριες γραμμές και ε, οικονομικές πολιτικές και πάλι λόγια, λόγια, lip service αυτά έρχονται και μας τα λένε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και πάλι για τον Google, για τις πέντε βασικές ε, προοπτικές του στόχου, ας πούμε και πώς συνδέεται αυτό με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο συμφωνώ αυτά που, που είπε ανησυχώ και εγώ το έχω ξαναπεί και ποιε είναι οι συνέπειες συμφωνώ. Σε σχέση με τον Έντουαρτ Σικλούνα, ευχαριστώ πολύ. Ενισχύουν αυτά που λέτε και αυτά που μας είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου όταν ήρθε εδώ να ε, παρουσιάσει την κατάσταση της Ελλάδας. θέμα δεν ήταν ε, ο ένας να κατηγορεί τον άλλον ή όλοι να κατηγορούν έναν. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι και όλοι υπέτοι και όλοι ένοχοι. Και όσοι είναι δακτυλοδεικτούμενοι δεν μπορούν να σωθούν αν δεν αναλαμβάνει ο καθένας τις ευθύνες του. Ο καθένας. Ε, και αν δεν λειτουργούν σωστά ε, τα θέματα της αλληλεγγύης και του συντονισμού. Και αυτό είναι ένας από τους πυλώνες οικονομικής διακυβέρνησης που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ως προαπαιτούμενο αν θέλουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο να είναι επιτυχία και όχι μια αλληλουχία εποπτείας και κυρώσεων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω το χρονοδιάγραμμα. Το σχέδιο έκθεσης θα υποβληθεί 14 Ιουνίου με Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών 21 Ιουνίου, συζήτηση των τροπολογιών στις 11 Ιουλίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή στις 12 Σεπτεμβρίου, με στόχο να περάσει από την Ολομέλεια στην η Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Ε, θα έχουμε χρόνο για να μελετήσουμε και να διερευνήσουμε τις ε, καλές ιδέες που συζητήσαμε. Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν στη συζήτηση. Το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διαταξία από σήμερα είναι το 8. Η εγγραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόκτηση νέων εμεριδίων στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη. Και εγώ την χάνει να είμαι εισηγήτρια. Η έκθεση είναι πολύ σύντομη και επί της ουσίας, διότι προτείνω να εγκρίνουμε την προτινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Συγκρότησης και Ανάπτυξης από 15 σε 30 δις ευρώ. Και στόχος αυτό είναι να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει και να αποκτήσει νέα μερίδια στο μετοχικό κεφάλαιο της Μπέρντα σε σχέση με το σημερινό μερίδιο της Ένωσης σε αυτό το κεφάλαιο και αυτό, για ποιο λόγο, διότι Η τράπεζα ανταποκρίνεται στις επιπτώσεις ε, της κρίσης και θεωρείται ότι υπήρξε σημαντικός αντίκτυπος ως αποτέλεσμα της κρίσης στον τομέα λειτουργίας της και γι' αυτό και θέλει να μπορέσει να συνεχίσει να απαλύνει τα επιπτώσεις της κρίσης και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θα την διευκολύνει να κάνει ακριβώς αυτό. Θεώρησα λοιπόν ότι ήταν καλή η σύσταση αυτή και τη συστήνω και στους συναδέλφους. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. No takers, right, well. Ωραία, λοιπόν, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 19 Απριλίου. Α, συγγνώμη. Σπέν, συγγνώμη. Ναι, να σου πω ότι έχουμε λοιπόν Προθεσμία υποβολή τροπολογιών 19 Απριλίου, εξέταση τη έκθεση 24 Μαου, ψηφοφορία στι 24 Μαΐου με στόχο να περάσει από τη δεύτερη ολομέλεια του Ιουνίου. Ο Σβέν, ναι, θέλω μόνο να πω μερικά πράγματα ε, και να πιστήσω την προσοχή σας αυτό. Φυσικά, όταν δει κανείς την ε, δημοσιονομική κρίση και την έλλειψη συνοχής, οικονομικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματικά χρειάζεται να έχουμε δομές τραπεζικές όπως η Bird και η ΕΤΕ. E Αλλά αν εξετάσουμε την συμπεριφορά τους, αν αξιολογήσουμε τη συμπεριφορά τους, θα πρέπει να δούμε ότι η δράση τους δεν συμφωνεί με τους κλιματικούς μας στόχους. Ε, ερευνούν, ας πούμε, δομές ε, στερεών καυσίμων στη Ρωσία, στο Καζακστάν, στη Ρωμανία, στην Σλοβενία, στη Μογγολία. Και το ερώτημα είναι, πρέπει να βάλουμε και άλλα χρήματα σε αυτή τη δομή χωρίς να αμφισβητούμε τη συνέπεια της πολιτικής τους, τη συνοχή των πολιτικών τους με τους γενικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των στόχων 2020. Ε, Πιστεύω πως ε, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να θίξει τα θέματα αυτά και για να εξασφαλίσει ότι επιπλέον χρήματα, τα επιπλέον χρήματα δεν θα χρησιμοποιηθούν ε, ώστε να προχωρήσουν σε μια κατεύθυνση κατά των γενικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελικά. Αντίθετη. Βέβαια έχουμε μια διπλή δομή. Έχουμε την BERD και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Γιατί έχουμε δύο διαφορετικές τράπεζες. Ξέρω πως ε, είναι διαφορετική η δομή συμμετοχής, διαφορετικές χώρες καλύπτονται, αλλά υπάρχουν και πολλές επικαλύψεις και αυτό θα πρέπει να το ε, αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό στην έκθεση αυτή θα κάνουμε τροπολογίες ώστε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις και να πετύχουμε η Μπέρντ να διαλυθεί μέχρι το 2015 και να δημιουργηθεί μια δομή μέσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που να είναι πιο αποτελεσματική και τελικά και πιο δημοκρατική. Γιατί εφόσον έχουμε περισσότερη δυνατότητα επιρροή στην, στην ε, ε, ΕΤΕ παρά στην ΜΠΕΡΤΑ. Ε, νομίζω πως αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουμε και χρειαζόμαστε περισσότερες δημόσιες τράπεζες, κρατικές τράπεζες για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις σωστές επενδύσεις που να είναι όμως βιώσιμες και να μην συνεχίσουμε με τη διπλή δομή δύο διαφορετικών τραπεζών που να λειτουργούν βασικά στην ίδια κατεύθυνση. Και θα το εκτιμούσα αν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε μια γραμμή που να ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε εδώ κάποιον από την Κομισιόν που ίσως να μπορεί να μας ε, ενημερώσει κάπως περισσότερο. Κύριε ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να συνταχθώ με την ε, τελευταία σας σύσταση που λέει πως η πρόταση δεν είναι πολύ επίμαχη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Εγώ κοίταξα την ιστορία αυτής της τράπεζας γιατί η Τσεχοσλοβακία και η Τσεχία μετά χρησιμοποίησε κάποιες επενδύσεις σε αυτές τις τράπεζες στις αρχές της δεκαετίας του 90 και αναζητούσε την απάντηση πόσο επιτυχής ήταν η ΕΤΑ και γύρω στο 90% και ίσως έτσι απαντάμε στον κύριο Γκίγκολντ σχεδόν 90% των επενδύσεων της ΕΤΑ στην Τσεχοσλοβακία αφορούσε ξένες επενδύσεις από την Δύση. Οπότε ίσως να ήταν αυτός ένας τρόπος να βοηθηθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, στις χώρες που αναφέρατε. Το ένα είναι αυτό. Προσωπικά εγώ Βλέπω λίγο επιφυλακτικά το, το ότι σε καιρούς στην εποχή δημοσιονομικών πραγματο, πραγματικοτήτων μια αύξηση 50% είναι τεράστια και πρέπει να λάβουμε υπόψη μήπως ε, παρά είναι, παραπάει. Το επόμενο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το μέλλον. Οι μελλοντικέ επενδύσεις, ε, επενδύσεις με συγχωρείτε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και Ανάπτυξης και το πώς τα εθνικά κοινοβούλια θα εμπλακούν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων για το πού και ποιες επενδύσεις θα γίνουν. <coughs> Αυτά τα τρία σύντομα σχόλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παθαίνουμε τώρα στην Κομισιόν. Βεβαίω, για αυτά τα ζητήματα λέμε πως δεν υπάρχουν επιπτώσεις στον προπολογισμό, γιατί βεβαίω τα χρήματα είναι απαιτητά αντί για καταβληθέντα. Αλλά καμιά φορά τα, απαιτούν κιόλα. Κάποια στιγμή κάποιος θα τα απαιτήσει κιόλα. Βίκυ, ήθελες να πεις κάτι. Ο Σβέν είπε για τις δύο τράπεζες. Εγώ καταλαβαίνω πως είναι τελείως διαφορετική η μετοχική δομή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση δεν έχει μόνο Ευρωπαίους μετόχους. Μάλιστα. Άλλες ερωτήσεις για προς την Κομισιόν. Κοιτάξτε για μένα. Ε, για να καταλάβω, θέλω να καταλάβω ακριβώς πώς δικαιολογείται ε, με τους ευρωπαϊκούς ε, στόχους, τους κλιματικούς. Ε, πηγαίνουμε για ένα μείον 8% στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ταυτόχρονα έχουμε αυτή την τράπεζα να επενδύει σε κάτι που αντιβαίνει αυτούς τους στόχους. Θέλω μία απάντηση. Thank you very much. already mentioned Argentina... Μια που αναφέρατε ήδη την Αργεντίνα, την Αργεντινή. Την Αργεντινή. Ξέρετε πώς σταμάτησε τις ε, πληρωμές της στην ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οπότε καμιά φορά, όπως είπα, είναι απαιτητά αυτά τα κονδύλια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω πρώτα απ' όλα για την αύξηση, το μέγεθος της αύξησης του κεφαλαίου. Ε, οι διοικητέ αποφάσισαν την αύξηση αυτή και αυτό προκύπτει από τις ανάγκες της κρίσης και για να μπορέσουν βεβαίως να ανταποκριθούν και στον, ε, ε, στην επάρκεια την κεφαλαϊκή της τράπεζας και βεβαίως να διατηρήσουν ε, την αξιολόγησή τους που είναι 3α. Οπότε θα υπάρξει αυτή η αύξηση του κεφαλαίου και θα αναθεωρηθεί στο τέλος της περίοδου για να δούμε αν χρειαστεί να διατηρηθεί ή σε κάποιο κεφάλαιο θα επιστραφεί. Επίσης, όπως σωστά είπατε, μιλάμε και για το απαιτητό και για το καταβληθέν κεφάλαιο. Το απαιτητό κεφάλαιο δεν, απαιτεί κάποια εκταμίευση, ε, καθώς μιλάμε για μετατροπή αποθεματικών. Επίσης είπατε πως το απαιτητό κεφάλαιο καμιά φορά απαιτείται κιόλα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο σε καμία από τις δύο τράπεζες το είναι περισσότερο θεωρητικό το ζήτημα. για την αλληλεπικάλυψη μεταξύ των δύο τραπεζών από δύο πράγματα. Τα δύο αυτά, οι δύο αυτές τράπεζες δημιουργήθηκαν σε διαφορετικό χρόνο για να ανταποκριθούν σε διαφορετικές ανάγκες. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ναι, κυρίως ε, αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση 90% των δραστηριοτήτων της είναι εντός των κρατών μελών και μιλάμε κυρίως για επενδύσεις σε έργα υποδομής κτλ ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και ανάπτυξη έγινε για να υποστηρίξει τις ανατολικές χώρες για να μεταβούν σε μια οικονομία της αγοράς και κυρίως πράγματι ενισχύει τον ιδιωτικό τομέα. Διαφορετικές οι πολιτικές λοιπόν. Και άλλα σωστά επισημάνατε πως υπάρχουν κάποιες αλληλεπικαλύψεις. Ε, Γι' αυτό, παραδείγματος χάρη, ε, υπέγραψαν ε, οι δύο τράπεζες ένα μνημόνιο για να είναι πιο σωστή η συνεργασία τους και να μην υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους. Τώρα, για το κλίμα δεν είμαι εγώ ειδικό αλλά νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης ε, και Ανασυγκρότηση έχει αυξήσει πάρα πολύ τις επενδύσεις της ε, σε παρόμοια έργα και ε, ενεργειακή αποδοτικότητα κτλ. Δεν είμαι σίγουρος το αν η πολιτική αυτή είναι κατά των κλιματικών στόχων της Ένωσης. Νομίζω πως υπάρχει μια σαφής ε, προσπάθεια αύξησης των επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα. Again, I mean, I'm, I'm very grateful that, that you are, let's say, um, have a very uh, shortened... Οπότε, ε, Κοιτάξτε, μέχρι το τέλος ε, του έτους ούτως ή άλλως ε, θα πρέπει να υπάρξει αυτή η αύξηση του κεφαλαίου. Σας ευχαριστώ, δεν ζητάει το λόγο και μια που έχουμε χρόνο. Πολύ γρήγορα, πάρα πολύ σύντομα. Το ζήτημα είναι το εξή. Καταρχάς σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν έχω ενοποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Καλό είναι που αυξάνετε τις πράσινες επενδύσεις και καλό είναι και για τη σύγκληση και ό,τι άλλο θέλετε. Αν θέλετε όμως, αν μέχρι το 2015 50 μάλλον, πρέπει να φτάσουμε στο μείον 80 και μείον 90%. Τι θα γίνει με ε, τις ρηπαίνουσες τεχνολογίες ε, ε καυσίμων οι θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, αν γίνουν εκεί επενδύσεις για να αποδώσουν και να αποσβεστούν, είναι μακροχρόνιες, μακροπρόθεσμες και συγκρούνται με τους στόχους για το κλίμα. Ίσως θα μπορούσατε να μας απαντήσετε γραπτός, γιατί για μένα είναι η προϋπόθεση για μια υπερψήφιση των πρασίνων. Δημοκρατικά ε, αποφασισμένες ε, λύσεις και στόχοι είναι αυτά. Η Πρόεδρος. Αν έχετε κάποια σχόλια παρακαλώ ε, να τα στείλετε γραπτός. Γιατί παραδέχτηκε ο Επίτροπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν είναι ειδικό σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής. Η Βίκη Φόρτ. Ναι, ε, σε σχέση με αυτό που είπε ο Σβέν για τη διαφάνεια. Είναι πολύ ωραίο να είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν έχουμε Απαντήσει για τις ε, ε, πολιτικές επενδύσεων και κρίμα που δεν είναι εδώ αρμόδιος. Είναι πολλά τα λεφτά και πρέπει να μας ενημερώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, τα υπάρχοντα δάνεια, πώς αποδίδουν, αν αποδίδουν, πού επενδύονται τα χρήματα αυτά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξης. Χρειάζεται πάρα πολύ υποδομή, ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, όχι μόνο η παραδοσιακή επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και επέκεινα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε γιατί χρειάζεται αυτή η κλίση κεφαλαίου κτλ. Στείλτε μας και με email πληροφόρηση. Θα μας βοηθούσε αυτή πολύ. Ευχαριστώ. Astrid. Η Άστριτ Λούλινγκ. Ε, κυρία Πρόεδρε, εγώ έχω μια ερώτηση αρχής. Ποιος είναι ακόμα λόγος ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης συστάθηκε για να εξασφαλιστεί η μετάβαση των κομμουνιστικών κρατών προς ένα δημοκρατικό πολίτευμα και μια οικονομία της αγοράς. Ολοκληρώθηκε αυτή η μετάβαση. Είναι και πλήρη μέλη στο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές οι χώρες. Καλά είναι αυτά που ακούμε, συνεργάζονται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η BERD, αλλά κάποια στιγμή να αναρωτηθούμε τι θέλουμε, ακόμα τι χρειαζόμαστε αυτή την τράπεζα. Και σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις της. Κατά την άποψή μου αυτό θα πρέπει να γίνεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Um, uh, Sven, if you're going to speak, do it on Sven, ε, θα τα αν θε να μιλήσεις πρέπει να το κάνεις με μικρόφωνο. Δεν σε ακούμε αυτά που λε. Πολλέ ερωτήσεις έκανες. Εγώ από ό,τι κατάλαβα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα συγκρότηση και Ανάπτυξης θέλει να επεκτείνει τον τομέα δραστηριοτήτων της περισσότερο προ τη Μέση Ανατολή. Αυτό έχω αντιληφθεί εγώ. Αλλά ίσω να μπορούσαμε να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να τη ζητήσουμε μάλλον απαντήσει σε όλε τι ερωτήσει που έγιναν και αν χρειαστεί Μπορεί να ρωτήσουμε και την ίδια την τράπεζα ανασυγκρότηση και ανάπτυξη. Αν έχουν πιο σαφέ όραμα, γιατί χρειάζονται επιπλέον ε, χρηματοδότηση και πού θα δαπανηθεί αυτή. Και η επέκτασή τους προς τα πού είναι γεωγραφικά. Τι τομεί θα καλύπτονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας έδωσα ήδη το χρονοδιάγραμμα, αλλά δεν έχουμε διάφορα. Οπότε η επόμενη συνεδρίασή μας είναι την 3η 19 Απριλίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Λήξεις.